Καλησπέρα σας. Θα, ήθελα να ξεκινήσουμε παρακαλώ τη συνεδρίασή μας. Βρισκόμαστε στο σημείο 9, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για το Συντονισμό των Ευρωπαϊκών Πολιτικών, τις ε, πτυχέ απασχόληση και τι κοινωνικέ πτυχέ στην ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη του 2017. Πρώτη εξέταση. Θα δώσω το λόγο στην εισηγητριά μας, την κυρία Γιάννα Τούμ. Κυρία Ριμπέιρο, συγγνώμη. Ε, θα μιλήσω πορτογαλικά. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα στη φάση αυτή να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας με όλο το σεβασμό που τρέφω προς την ε, Πρόεδρο, του συναδέλφους και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να πω ότι ε, είμαστε μόνο οι σκιώδεις Δεν χρειαζόμαστε κανονική δημόσια συνεδρίαση για να συνομιλήσουμε. Πραγματικά δεν έχει νόημα. Πάμε να πιούμε ένα καφέ εις και ό,τι συγγητές και να το πούμε. Δεν χρειάζεται τώρα να εξηγούμε από την αρχή τις θέση μας, αφού δεν έχουμε άλλους συναδέλφους. Μπορούμε να το κάνουμε και αλλού αυτό. Όχι σε μια συνεδρίαση που είμαστε τρεις και ο Κούκος. Δεν ξέρω, ίσως έχει νόημα να αναβάλουμε τη συζήτηση. Βέβαια, επαφή με στην Πρόεδρο. Αν η αποφασίσει η Πρόεδρος να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση, πολύ ευχαρίστως να μιλήσω για το σημείο αυτό. Τηρώντας αυστηρά τις ε, αρμοδιότητες και τα καθήκοντά μου. Αλλά ό,τι πει η Πρόεδρος. Any other comments, reactions? υπάρχουν άλλα σχόλια, ε, παρατηρήσεις ε, για την πρόταση της κυρίας Ριμπέρο. Για να το. Να πω, μια και βρεθήκαμε, θα σου πω και εγώ δύο λόγια για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Το πακέτο ε, δημοσιεύθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2016 και η λόγω γνωμοδότηση δίνει τη γνώμη μας για τις κοινωνικές πτυχές και τις πτυχές απασχόλησης στην ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης για το 2017. Είχαμε σχετικά πρόσφατα χαρμόσυνες ειδήσει. Φαίνεται ότι αρχίζει και ανακάμπτει η ευρωπαϊκή οικονομία. Βέβαια, θα πρέπει να δημιουργηθούν και θέσει απασχόληση. Το 2013-2016 δημιουργήθηκαν 8 εκατομμύρια νέε θέσει απασχόληση. Και από 8,5% το 2018 έχουμε. Ε, το 2016 είχαμε το 8,5% ε, ποσοστό έχει μειωθεί και το ποσοστό απασχόληση αντίθετα είναι 71,71%. Πολύ καλύτερα από το 2008 που ήταν 70,3% το ποσοστό απασχόληση. Βέβαια, ο στόχος ε, της Ευρώπης 2020 ε, είναι 75% ο στόχος του ποσοστού απασχόληση. και ε, βλέποντας τα σημερινά νούμερα μάλλον απεσιόδοξη είμαι για το κατά πόσο θα υλοποιήσουμε αυτό το στόχο του 75% απασχόληση. Τώρα, ω προς το θέμα αυτό, θα πρέπει να ενισχύσουμε καταρχήν την εφαρμογή της ε, εγγύηση για την νεολαία. Να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τα μεμονωμένα ε, ειδικά μέτρα για τους μακροχρόνια ανέργους. Επίσης, την αντιστοίχηση ε, δεξιοτήτων και προσόντων με τις ανάγκες για νέες θέσεις ή τις ανάγκες της αγοράς. Επίσης, το θέμα της κατάρτισης και της αμοιβέ αναγνώρισης των προσόντων και δεξιοτήτων είναι πολύ σημαντικά αυτά. Και να μην ξεχνούμε και το ρόλο των επενδύσεων, ιδιαίτερα στις ε, ψηφιακές δεξιότητες. Και μάλιστα από επιθεωρήσεις εργασίας ή από άλλους αντίστοιχους φορείς, στον χώρο που δεν έχουν τέτοιες ε, επιθεωρήσεις εργασίας, έγινε μια προσπάθεια να θεσπιστούν κάποια μέτρα για να μπορέσουν να προσαρμοστούν καλύτερα στις ε, ανάγκες της παγκόσμιας οικονομίας οι εργαζόμενοι. Επίση, θα πρέπει να αυξηθούν τα κίνητρα για του εργαζόμενου και τα φορολογικά συστήματα μπορούν να συμβάλλουν στην καταπολέμηση των ανισοτήτων του εισοδηματικών. Επίση, να δώσουμε έμφαση σε ε, δραστήριες πολιτικές υπέρ τη απασχόλησης σε στενή συνεργασία με τους ε, κοινωνικού εταίρους. Επίση αναγνωρίζω ότι το ποσοστό ανθρώπων που κινδυνεύουν από ένδια και αποκλεισμό είναι υψηλό. Το 2015 στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 190 περίπου εκατομμύρια οι συνάνθρωποι μας ε, σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και ένδια. Θα πρέπει να μειώσουμε αυτές τις ανισότητες γιατί υπονομεύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η δημιουργία θέσεων απασχόληση είναι αποτελεσματικό μηχανισμό για την καταπολέμηση τη ένδυα και να μην αγνοούμε και το ρόλο των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεδομένη και τη γύραση του ευρωπαϊκού πληθυσμού, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνική πρόνοια και ανάπτυξη στρατηγικών για να παραμείνουν ε, πιο ηλικιωμένοι, ε, ενεργοί στην κοινωνία μας. Και τα ευρωπαϊκά ταμεία μπορούν να διευκολύνουν καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, να αυξήσουν τις επενδύσεις και να τονώσουν την επιχειρηματικότητα. Επίσης να, ε, να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία με βάση και τις ειδικές συστάσεις αναχώρα. Και πιστεύω επίσης στο πλαίσιο της καταπολέμησης της φτώχειας τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κάποιες ελάχιστες κοινωνικές προδιαγραφές. Και ευελπιστώ ότι θα με στηρίξουν και οι συνάδελφοι στις προτάσεις μου. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και περιμένω τα σχόλιά σας και με ιδιαίτερη χαρά θα λάβω μερικά τουλάχιστον από αυτά υπόψη. Εμεί ευχαριστούμε τώρα για να σχολιάσουμε την ε, προηγούμενη πρόταση τη κυρία Ζεμπέρα. Πρέπει να πούμε ότι πάντοτε υπάρχει αυτό το πρόβλημα σχεδόν σε όλες τις επιτροπές. Έτσι γίνεται τις πέμπτες το απόγευμα. Τώρα είμαστε πεθαμένοι στην κούραση, σκεφτόμαστε τα Χριστούγεννα, οπότε χρειάζεται να επιβιώσουμε λίγες μέρες παραπάνω ε, και για το Στρασβούργο όσον αφορά την ψηφοφορία. Τι να σας πω. Δεν, δεν, δεν, δεν φτάνει αυτό. Αλλά υπάρχει τελικά κάποιο περιθώριο ελιγμών. Και άρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα ξαπούμε κάποια στιγμή αργότερα. Είναι προβληματική η κατάσταση και με τις αίθουσες ε, και η μέση διάταξη είναι αυτή που είναι και η κυρία Τούν μας τα είπε. Και πολλοί παρακολουθούν την συνεδρίαση, αλλά από μακριά, όχι από μέσα από την αίθουσα. Με άλλες μεθόδους μας ακούν. Τέλος πάντων. Αυτό το είπα για την πρότασή σας. Για πέστε μας για την έκθεση, κυρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αφού αυτή είναι απόφαση την οποία αναπαντή, θα μιλήσω σχέση με αυτό το ε, ζήτημα και ε, δείχνοντα σεβασμό και σε εσά ω πρόεδρο και απέναντι στην κυρία Γιάννα Τόμα, η οποία έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά σε σχέση με αυτό το ζήτημα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τη συνάδελφο Γιαννατούν για το έκθεση που μας παρουσίασε και η οποία βέβαια σηματοδοτεί την έναρξη των συζητήσεών μας ε, σε σχέση δηλαδή με το τι θέλουμε να έχουμε στο μέλλον στην Ευρώπη, ειδικότερα σε σχέση με τα κοινωνικά ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να κάνω κάποιες προτάσεις σε ό,τι αφορά αυτή την πρόταση και τις οποίες βέβαια θα εμποβάλω και γραπτώ στη συνέχεια. Καταρχήν, θα ήθελα να τονίσω ότι θα πρέπει να νομιμοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Και δεν θα πρέπει δηλαδή να επαναληφθούν καταστάσει όπω αυτέ που είχαμε φέτο, όπου για παράδειγμα η Πορτογαλία και η Ισπανία ενδεχομένως να έμπαιναν σε μια διαδικασία τελικά επιβολής κυρώσεων χωρίς να έχει καταλάβει ποτέ ακριβώς κανείς τι έχει ε, συνέβη. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην διαδικασία της νομιμοποίησης αυτού του Ευρωπαϊκού Εξάμενου. Από εκεί και μετά ε, βρισκόμαστε ακόμα σε μια οικονομική κατάσταση η οποία παραμένει εύθραυστη. Οπότε θα πρέπει να εστιάσουμε και να παραμείνουμε εστιασμένοι σε δύο βασικούς στόχους. Δηλαδή να αυξήσουμε την οικονομική ανάπτυξη και τι εργασίας και αυτό σημαίνει δηλαδή να προβούμε στις επενδύσεις, να ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις, να προβούμε σε βιώσιμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να ε, προβούμε και σε υπεύθυνες σχετικές περιβαλλοντικές ε, πολιτικές. Ε, ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη συνέχιση της υψηλή ποιότητας του κοινωνικού μοντέλου της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση οι τρεις πυλώνε που μόλις τώρα ανέφερα ε, ε, δεν θα εφαρμοστούν με τον τρόπο που πρέπει και θα αμφισβητηθεί σύντομα το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτή της έφραση της οικονομική ανάπτυξη που βιώνουμε δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για δύο εκατομμύρια επιχειρήσει που απασχολούν γύρω στο 7% των εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν με αυτόν τον ε, τρόπο δίνουμε ε, και καταδεικνύουμε ακριβώ την ανθεκτικότητα που έδειξαν αυτέ οι επιχειρήσει σε ό,τι ακριβώ αφορά τη διατήρηση της ποιότητα του κοινωνικού μοντέλου τη Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε τι προποθέσει έτσι ώστε οι επιχειρήσει μα να συνεχίσουν ε, να αυξάνουν την δυνατότητα παραγωγής τους. Και όταν αναφερόμαστε σε παραγωγικότητα, συχνά ε, εννοούμε ε, τις ε, ώρες εργασίας αναπαραγωμένο προϊόν. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με ειδικότερα με αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά δηλαδή, την καλύτερη αξιοποίηση όλων των πόρων συμπεριλαμβανομένων και αυτών του ανθρωπίνου δυναμικού. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αυξήσουμε την ε, ε, αποδοτικότητα των επιχειρήσεών μας και ε, κατά συνέπεια και την παραγωγικότητά τους. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε αυτή την αποδοτικότητα θα πρέπει να κάνουμε τις κατάλληλες επενδύσεις στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση και θα πρέπει να γίνει κατάλληλος διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους, ε, τις, τους εκπαιδευτικούς φορείς, και φυσικά όταν αναφέρουμε στους κοινωνικού εταίρους αναφέρουμε και στις συνδικαλιστικές οργανώσεις αλλά αναφέρουμε και στις δημόσιες επιχειρήσεις και σε άλλους συναρμόδιους φορέ. Όλοι λοιπόν αυτοί θα πρέπει να ε, συνεχίσουν τις προσπάθειες που κάνουν σε όλα τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να καλυφθούν πραγματικά οι ανάγκες που έχουν οι επιχειρήσεις σε σχέση με την αύξηση της παραγωγικότητας. Και δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι ε, το 25% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση έρευνα του ΩΣΑ διαπιστώνει ότι η, ο επίπεδο των δεξιοτήτων τους ε, δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που θα ήθελαν για τις ανάγκες της συγκεκριμένης επιχείρησης. Δεν λέμε δηλαδή ότι είναι υπερβολικά χαμηλές οι δεξιότητες τους, απλώς αναφέρουν εν λόγω εργαζόμενοι ότι ε, δεν ανταποκρίνονται στο επίπεδο που θα είναι το πλέον χρήσιμο για την επιχείρηση. Άρα λοιπόν ε, θα πρέπει να παραμείνουμε εστιασμένοι στους βασικούς μας στόχους μεταξύ αυτών δηλαδή και στην αύξηση των θέσεων εργασίας ε, και βρισκόμαστε πραγματικά σε καλό δρόμο, βρισκόμαστε σε μια σε ένα ποσοστό απασχόληση τάξη του 71,5% οπότε πραγματικά ενδεχομένω να είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε ε, τις ε, προτεραιότητες ε, της του 2020 αλλά για να το πράξουμε θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το όραμά μας θα πρέπει να παραμείνει ένα όραμα συνοχής που σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε έμβαση στις εξόχως απόκεντρε ε, περιοχές και γενικότερα στις ε, μειονεκτούσες ε, περιοχές. Ε, κλείνοντας... Ε, να πω ότι έχει διαπιστωθεί κάτι και σε επίπεδο δηλαδή ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ακριβώς αυτές τις τρεις, την ισορροπία ανάμεσα στους και οικονομικούς επιλώνες και ε, στο κοινωνικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα πρέπει δηλαδή να έχουμε πάντα κατά νου ότι όλα αυτά εξυπηρετούν τελικά το συμφέρον των πολιτών μας και κατά συνέπεια και τον Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ε, θα δώσει ένα θετικό ένωσμα στην κοινωνική ανάπτυξη της Ευρώπης. Οπότε θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα διατηρηθεί η εν λόγω ισορροπία και ακριβώ οι δικέ μα ε, γραπτέ ε, τροπολογίε θα κινηθούν προ αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να διασφαλίσουν αυτή την ισορροπία και μέσα στο κείμενο τη έκθεση. Ευχαριστώ. Ε, thank you. Σας ευχαριστούμε κύριε Ριμπέιρο. Η Μαρία Ρενά είναι η σκιώδη συγγετρία των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Μήπως την αντικαθιστάτε εσείς κύριε Πυρίνσκι. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, είπατε στην αρχή ότι η σε αυτή είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία εξέτασης ε, του σχεδίου έκθεσης. Θα ακολουθήσουν οι τροπολογίες, οπότε θα ακολουθήσει και συζήτηση για την εξέταση των τροπολογιών. Γιατί και εγώ συμφωνώ με την κυρία Ριβέρο δεν μπορεί να γίνει εδώ ουσιαστική συζήτηση. Γιατί περισσότεροι λείπουν. Και εμείς από σεβασμό προς την εισηγήτρια και το έργο της ε, δεχτήκαμε να μας κάνει την παρουσίαση της έκθεσης, αλλά το θέμα της αιτήσια επισκόπησης για την ανάπτυξη και ιδιαίτερα των κοινωνικών πτυχών και των πτυχών απασχόλησης ε, της αυτή αυτής επισκόπησης είναι ε, θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων της Επιτροπής και των αρμοδιοτήτων και υποχρεούμεθα να προβούμε σε ευρυθή και σοβαρή εξέταση του θέματος και της σχετικής έκθεσης της κυρίας Τούμ. Τώρα ως προς την έκθεση καθ' αυτή. Θεωρώ ότι κάνει μια σφαιρική προσέγγιση του θέματος υπό το πρίσμα των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας και περιλαμβάνει τα βασικά θέματα που μας ενδιαφέρουν. Ίσως θα, αυτό που θα μπορούσα να προτείνω θα ήταν να κατεβάσουμε λίγο τους υπεραισιόδοξους τόνους της έκθεσης. Γιατί στηρίζεται στα στοιχεία περιμείωσης της ανεργίας και αναφέρει τα πολλά αριθμα μέτρα που ελήφθησαν. Όχι ότι αυτά θα πρέπει να τα αγνοούμε, αλλά ίσως θα πρέπει να εγγύψουμε πιο διεξοδικά και πιο σχολαστικά στις δράσεις που λαμβάνονται πίσω από τα φαινομενικά τουλάχιστον θετικά στοιχεία και τη βελτίωσή τους. Σε ό,τι φορά την κατάσταση στην απασχόληση, για παράδειγμα, σε πολλές περιπτώσεις η μείωση των επίσημων των επίσημα ανέργων Ε, σχετίζεται με την αύξηση κάποιων επισφαλών μορφών απασχόλησης ή μορφών ψεύτο αυτοαπασχόλησης. Οπότε, αν στηριχθούμε αποκλειστικά και μόνο στην φαινομενική βελτίωση του ποσοστού ενεργείας που δείχνουν τα στοιχεία εκ αυτό δεν αρκεί. Αναγνωρίζουμε με τη μείωση αυτή της ενεργείας, αλλά θα πρέπει να παραμερίζουμε τους παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή τη φαινομενική μείωση. Και η βασική ανησυχία που α, σήμερα ε, ασθενιζόμαστε με την εισηγήτρια είναι ότι σε τελική ανάλυση, ακόμη και η οικονομική ανάπτυξη είναι ε, απειροελάχιστη, περιθωριακή και δεν οδήγησε σε αύξηση της, της ζήτησης, ε, σε τόνωση της οικονομίας ή σε αύξηση των θέσεων απασχόλησης ή τουλάχιστον με τρόπο που να επηρεάσει ε, αισθητά την κατάσταση. Συμφωνώ ε, με την έκκληση να εγγύψουμε στο θέμα της αδήλωτης εργασίας, παράγραφος 8, και να ζητούμε από τα κράτη-μέλη να προβλέψουν είτε επιθεωρήσεις εργασίας είτε αντίστοιχους φορείς και να τους εφοδιάσουμε τους απαραίτητους πόρους. Κατέθεσα και μία τροπολογία κάπως πιο φιλόδοξη που αναφέρει και την σημασία των πλατφορμών για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Έχει ληφθεί ήδη απόφαση για την σύσταση αυτής της πλατφόρμας και περιλαμβάνεται και στο πρόγραμμα εργασιών. Έχει ήδη οργανώσει ε, η πλατφόρμα αυτή ένα σεμινάριο για τους διάφορους δείκτες που λαμβάνονται υπόψη. Ας το αναφέρουμε λοιπόν και αυτό. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη του έργου της πλατφόρμας και θα μπορούσαμε αυτό να το αναγνωρίσουμε στο κείμενο, ενθαρρύνοντας περαιτέρω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνδράμει ακόμη περισσότερο την σχετική πλατφόρμα με τις δικές της δραστηριότητες. Προς το παρόν ε, αυτά. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω. χρειαζόμαστε εκτενή συζήτηση, γιατί είναι σοβαρά τα θέματα. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε και αυτά που επισήμανε η κυρία Ριμπέιρο. Έχουμε κάποιες χώρες που είτε εφαρμόζουν ακόμη μνημόνια, είτε μόλις έχουν, τα έχουν ξεπεράσει. Και στις χώρες αυτές ε, τα εισοδήματα είναι πολύ χαμηλά, τα συστήματα κοινωνικής προστασίας ε, έχουν συρρυκνωθεί και επιπλέον οι χώρες αυτές υπόκεινται σε μέτρα που δεν τους επιτρέπει να αντιμετωπίσουν τις σοβαρές προκλήσεις που έχουν ενώπιον τους. Και δίνεται η εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αφουγκράζεται επαρκώς τις ανάγκες των πολιτών, ούτε επικεντρώνεται στις ουσιαστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές οι χώρες. Επίσης, η μνήμα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Αναφέρεται ότι το Ταμείο αυτό συνέβαλε στη σύσφυξη της ε, συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, δεν τεκμηριώνεται με στοιχεία αυτή η δήλωση. Στην παράγραφο 12 αναφέρουμε ότι το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων επιτρέπει τη βελτίωση της ε, οικονομικής συνοχής των κρατών μελών. Ενώ τα στοιχεία μας δείχνουν ότι το αντίθετο κάνει το ΕΦΣΥ. Γιατί οι περισσότερες επενδύσεις γίνονται ακριβώς σε χώρες που ήδη έχουν υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης. Ενώ στις υπόλοιπες χώρες δεν γίνονται σημαντικές επενδύσεις. Το 60% των επενδύσεων πηγαίνουν στις 5% πλέον ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πολλές φορές το συζητήσαμε αυτό για το πώς λειτουργούν οι επενδυτικές τράπεζες και το ΕΦΣΥ και δημιουργούν μεγάλες προκλήσεις εν ώψη και της δεύτερης φάσης του σχεδίου Juncker, του επενδυτικού σχεδίου του Juncker. Αυτά είναι κάποια γενικά στοιχεία για την ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη για το 2017, αλλά θα πρέπει να ακολουθήσει πολύ πιο ευρυθή συζήτηση. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Πριν δώσουμε το λόγο στην κυρία Τρεμπίνσκη. Τρεμπέσιους, τρεμπέσιους. Σωστότερα. Πρέπει να σας πω ότι η άποψή μου ταυτίζεται με τη δική σας, κύριε Πυρίνσκη. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα, αλλά, αλλά Ούτω ή άλλω. Σα ενημερώνω ότι την επόμενη εβδομάδα, που είναι η τελευταία σύνοδο του Στρασβούργου έχουμε μια κοινή συνεδρία Οικονομικής Επιτροπής και απασχόλησης όσον αφορά αυτήν την ε, έρευνα τελευταια συνοδο του στρασβουργου εχουμε μια κοινη συνεδρια οικονομική επιτροπης και όσον αφορά την ερευνα ετησιας ανάπτυξη. οχι οσον αφορα ε, την έκθεση εκθεση τέλο πάντων για τις προειδοποίησεις στις 12 ε, Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο. Δεν λέω ότι έτσι μπαλώνονται όλα αλλά δίνετε μια δεύτερη ευκαιρία. Ελπίζω ότι δεν περάσετε τη βράδυ των Χριστουγέννων μέσα στην πολιτική ομάδα για να μπορέσετε να συμμετάσχετε. Αλλά τέλος πάντων. Ε, καμιά φορά. Δύσκολο να κανονίσουμε για συνεδριάσεις με τόσο κόσμο όπως ε, θέλετε. Κυρία Τρεμπέσιο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, Καθώ ε, τοποθετήθηκαν όλοι σε σχέση με αυτό το ζήτημα του Ευρωπαϊκού Εξαμένου, θα ήθελα να τοποθετηθώ κι εγώ. Ε, δεν είναι ευθύνη της ε, Προέδρου το πόσοι ε, συμμετέχουν σε αυτές τις συνεδριάσεις. Η πατία, δηλαδή εξαρτάται από εμά τους ίδιους. Οπότε ίσως θα πρέπει να το πούμε και εμείς τους συναδέλφους μας κάποια στιγμή ότι και πέμπτη απόγευμα θα πρέπει να προσέρχονται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά όμως τη συγκεκριμένη έκθεση θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συναδελφό για την εξαιρετική ε, έκθεση, γιατί πραγματικά είναι πιο ισορροπημένη και πιο αντικειμενική σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Ε, για παράδειγμα, μα αρέσει το γεγονό ότι τονίζει την αρχή τη επικορικότητα και ότι δίνεται περισσότερη έμφαση στο ρόλο των εθνικών ε, κρατών μελών. γενικά σημειώνει μια ελαφρώς θετική εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης ε, και της αγοράς εργασίας, της απασχόλησης δηλαδή. Πράγματι είναι θετικό αυτό, αλλά δεν ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να επαναπαυθούμε. Πολλές ε, περιοχές δηλαδή αντιμετωπίζουν ακόμα σημαντικά προβλήματα και η λόγω ανάκαμψη δεν σημειώνεται στις πιο αδύναμες περιοχές. Ένα παράδειγμα για παράδειγμα είναι η Ιταλία, η οποία τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη και με ένα αβέβαιο πολιτικό μέλλον και δεν έχει ακόμα επιλύσει τις οικονομικές της ε, προκλήσεις. Ε, ε, δεν μπορούμε λοιπόν να θέτουμε πάνω αυτό το πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο κύριος Μάριο Ντράγκη θα επαναλάβει ή θα ζητήσει και πάλι τη διατήρηση του, ζητήματος, του προγράμματος εξαγορών του, αλλά αυτό δεν επιλύει τα προβλήματα και μάλιστα μειώνει, κρατάει χαμηλά επιτόκια. Οπότε ε, δεν θεωρούμε ότι θα βοηθήσει αυτή η διατήρηση ειδικότερα τις ε, πιο αδύναμες ε, χώρες οι οποίες ήδη υποφέρουν από αυτά τα επιτόκια. Από εκεί και μετά υπάρχουν για παράδειγμα τεράστια χρέη, συσσωρευμένα χρέη, για παράδειγμα δημόσια χρέη σε ορισμένα χώρα ε, όπως για παράδειγμα ε, στη Γαλλία και αλλού. Οπότε πραγματικά κάποια στιγμή η, Ευρωπαϊκή, η Ευρωζώνη θα πρέπει να διαλυθεί ούτως ώστε να αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες ε, τα διάφορα κράτη-μέλη και να έχουν και τις δυνατότητες που τους χορηγεί σε επίπεδο πολιτικής σε το δικό τους συνόμισμα. Και βέβαια με τα όσα συμβαίνουν σε επίπεδο δημοκρατικών αλλαγών θεωρώ πως τα προβλήματά μας στο μέλλον θα αυξηθούν και δεν θα μειωθούν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Τόμ για αυτό το πολύ καλό έγγραφο, δηλαδή μια πολύ καλή καλή βάση για την περαιτέρω συζήτηση και αναμένω με ενδιαφέρον τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Δεν έχουμε κάποιον από την ΕΚΟΕ. Η Τζιν Λάμπερτ προεδρεύει σε κάποια άλλη συνεδρίαση, δεν μπόρεσε να παραστεί. Επομένω, θα δώσω το λόγο στην κυρία Άγκυρ. Ορίστε. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μισό λεφτάκι, θέλω να ε, καθισκάσω πρώτα-πρώτα την κυρία Τρεμπέσου. Δεν τα πάει καλά η Ιταλία, αλλά τελικά είσαι το συνταγμά τη την Κυριακή. Οπότε νομίζω ότι είναι καλύτερο από ό,τι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί περάσαμε 78 χρόνια που υπερασπιζόμαστε με αυτό το Σύνταγμα την ε, αυτοκυριαρχία μας, την εθνική κυριαρχία δηλαδή και έτσι αντισταθήκαμε σε αυτή την ε, ε, αναθεώρηση που ήθελε η Ευρώπη στη στρεβλή να μας επιβάλλει. Οπότε δείξαμε ότι είμαστε όριμοι για κάποια κυβέρνηση σταθερή για μια καινούργια εποχή. Αυτά για να σας καθησυχάσω. Για να την ευχαριστήσω για την εισήγησή της αλλά διαβάζοντας μου προκύπτει το εξής ερώτημα. Μα στην ίδια Ήπειρο ζούμε. Και δεν βλέπω καμία ανάκαμψη στην Ευρώπη. Δεν βλέπω να έχουμε τίποτε εξελίξεις θετικές που να έχουμε αυτού του είδους τις ε, θέσεις απασχόλησης κατά εκατομμύρια που πρόκειται να, να καταφέρει η Ευρώπη να προετύχει τους, το, ε, τους στόχους του 2020 με ανεργία 25%. Τουλάχιστον λέω για την Ευρώπη όπου ζω εγώ. Και εδώ πέρα έχουμε ένα σωρό μέσα ευρωπαϊκά, τα, οποία υποτίθεται ότι είναι οι φορείς ε, αυτής της προόδου, οι γιούρες κλπ. για την ανταγωνιστικότητα και θα πρέπει να γίνουν κάποιες μελέτες επιπτώσεων για να δούμε ακριβώς ποια είναι τα αποτελέσματα από την υλοποίηση τέτοιων πολιτικών, εφαρμογή τέτοιων εργαλείων και μέσων. Οπότε φοβερή η αισιοδοξία σας και τι να σας πω, εγώ έχω να σας πω ότι υπάρχει ακόμα μεγάλη ανεργία, σας το λέω διστακτικά. Επομένω, νομίζω ότι έτσι κάπω αμαυρώνεται αυτή η ιδανική εικόνα την οποία έχετε περιγράψει. Πολύ θα ήθελα να ζούσα στην Ευρώπη που περιγράφεται. Δυστυχώ όμω, ζούμε σε κάποια Ευρώπη που είναι τελείω διαφορετική η πραγματικότητα. Στη δική μου Ευρώπη Έχουμε 122 εκατομμύρια που βρίσκονται από το όλη τη Είναι ένας στους τέσσερις, 122 εκατομμύρια ξεχάσαμε να τους εντάξουμε εδώ. Να τους αναφέρουμε δηλαδή στο κείμενο. Άρα δεν είναι δυνατόν να παίζουμε με τις στατιστικές, με αυτού του τα μακρο νούμερα. Εντάξει, ε, μεταξύ μας εδώ αλληλοσυγχαιρόμαστε. Παρά το ότι η κατάσταση είναι τόσο κρίσιμη σε πάρα πολλά κρατημέλη και έτσι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση μέχρι ότου οι, οι Βρυξέλλες θα σταματήσουν να κασκούν πολιτικές αντιφατικές χρειάζονται διαφορετικέ μεταρρυθμίσεις, ε, χρειάζονται καινούριε δημοσιονομικέ, ε, φορολογικέ πολιτικές, δουλειά, απασχόληση δηλαδή στην αγορά. Θέλουμε τα κράτη-μέλη να επενδύσουν στις επιχειρήσεις. Να υπάρξουν τέτοιου είδους μέσα για τους προπολογισμού, να υπάρχει κάποιο είδους ε, φορολογική εποπτεία και έτσι θα μπορέσει κάτι να κάνει η Ευρώπη. Γιατί και ο κόσμος και οι επιχειρήσεις ε, έχουν τσακιστεί από όλα αυτά τα φορολογικά βάρη. Δεν μπορεί να χρηματοδότηση η μικροεπιχείρηση. Μα τι να τα κάνουμε τα καινούργια μέσα για την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων. Τα κάνει αυτά και από την άλλη μεριά λέει στα κράτη-μέλη να ασκούν αυτές τις πολιτικές εναντίον των επιχειρήσεων που θα έπρεπε να χρηματοδοτούν. Πρόκειται για σχιζοφρενική πολιτική της λιτότητας. Οι φοροαπαλλαγές και η ανάπτυξη θα έπρεπε να πηγαίνουν μαζί. Αλλά θα πρέπει να δώσετε κάποιο είδου κίνητρα για να πάμε στην ανάπτυξη και να υπάρξει φορολογική υπευθυνότητα. Αλλιώς θα ξεπεράσουμε τα 120 εκατομμύρια. Θα πάνε στα 800 και τελικά θα είναι η πλειοψηφία στα κρατη Thank you. I'll give the floor to Ευχαριστώ κυρία Μπιζότο τώρα. Grazie. Ευχαριστώ. Εγώ συμφωνώ με αυτό το σχέδιο. Εκθέσεις μόνο στο σημείο που ε, λέει το, το πόσο ανησυχεί η συγκίτρια για την αυξανόμενη φτώχεια γιατί έχουμε όλες αυτές τις ε, συνταγές οι οποίες είναι άχρηστες και κυκλοφορούν εδώ στο κοινοβούλιο. Τι να σας πω. Και ε, λέμε τι γίνεται με την Ιταλία, έχουμε όλους αυτούς τους πρόσφυγες, έχουμε τόσα εκατομμύρια ευρώ 60 ε, δις δίνουμε όμως από την άλλη μεριά στην Τουρκία. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Συγγνώμη με την Eurostat. Μιλάμε για πάρα πολλά εκατομμύρια. 17 εκατομμύρια, όχι, διορθώνει. 117 εκατομμύρια. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στριμωγμένοι οικονομικά στην Ιταλία. 117. Και κάνουμε ακόμα μία έκθεση. Και έχουμε τόσες άλλες εκθέσεις, τόσα ψηφίσματα, ανακοινώσεις της Κομισιόν. Αλλά θα πρέπει να βρούμε το θάρρος και να αντιμετωπίσουμε, να λύσουμε τα προβλήματα, να βρούμε το θάρρος, να πούμε ποια είναι τα προβλήματα. Είναι ακριβώς αυτές οι ευρωπαϊκές οδηγίες είναι αυτό το ενιαίο νόμισμα, το οποίο τους φτωχοποιεί όλους. Το 2009 δεν έχω ακούσει ούτε μία συζήτηση που να αφορά το θέμα του ευρώ. Γιατί να μην κάτσουμε και να προβληματιστούμε μια ωρίτσα, μια ωρίτσα όσον αφορά το ευρώ, να το, αν δουλεύει δηλαδή το σύστημα. Γελάτε, γελάτε εσείς, αλλά είναι εκατομμύρια τα που δεν γελάνε καθόλου. Δεν σου δώσω κακή κατάσταση. Την Κυριακή όμως γελάσανε γιατί νίκησε η Ιταλία στο δημοψήφισμα. Απελευθερώθηκαν, Προφερθήκαμε από τον ε, Ρέντζι. Δεν θα πρέπει να υποτιμούμε το πρόβλημα. Αλλιώ η κατάσταση θα πηγαίνει στο χειρότερο. Άρα δεν είναι θέμα που προκαλεί γέλιο. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Μα λειτουργεί, αποδίδει το ευρώ. Τι μπορούμε να κάνουμε να κάτσουμε και να το σκεφτούμε. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι όπως τα λέτε στην έκθεση. Καλά, άλλο είναι ο εισηγητή, αλλά παρακαλώ να σκεφτείτε, να προβληματιστείτε μία μόνο ρίτσα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ που τόσε ώρε χάνονται από παράλογε συζητήσει. Τι έγινε αυτά τα τελευταία χρόνια, τι έγινε μετά τη θέσπιση του ευρώ είναι σε καλύτερη κατάσταση ή σε χειρότερη η Ευρωπαίοι. Thank you. Σας ευχαριστώ. Ε, μήπως έχουμε κάποιον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα θέλετε το λόγο για το θέμα. κυρία, ο Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συζήτηση και σημειώνει τα σχόλιά σας. Άλλα σχόλια προς το παρόν δεν πρόκειται να κάνουμε, γιατί την επόμενη Δευτέρα στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Παρουσία της Επιτρόπου Τάισεν η Επίτροπος ε, θα λάβει μέρος με πολύ χαρά στη συζήτηση μαζί σας και στην ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ η συγγετριά μας τώρα, η κυρία Γιάννα Τούμ. Θα προσπαθήσω να είμαι λακωνική. Στην αρχή της συζήτησης είχατε να αίσθηση ότι όλοι ήμασταν στην ίδια πολιτική ομάδα, ότι ήμασταν όλοι ιδεάτες και έβαλα κάποια, κάποιες λέξεις κλειδιά στην έκθεση και συμφωνώ μαζί σας ότι η εικόνα αυτή ελπίζω να μην αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι τα κοινωνικά θέματα δεν είναι τόσο σημαντικά ε, και γι' αυτό δεν ήρθαν, δεν μπήκαν στον κόπο να έρθουν συνεδρίε, απλώ να έχουν άλλες ε, υποχρεώσεις. Επίσης μιλήσαμε για τις επενδύσει, την οικονομική ανάκαμψη. Είπα ότι ήταν κάπω αισιόδοξα τα στοιχεία και συμφωνώ εν μέρη και με τα σχόλια των ε, Ιταλίδων συναδέλφων. Κάθε φορά που μιλάμε για κοινωνικά θέματα, στο σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, συνήθω παίρνουμε ε, τη μέση θερμοκρασία κατά κάποιο τρόπο των ασθενών στα νοσοκομεία. Μερικοί είναι σε καλύτερη κατάσταση, άλλοι σε χειρότερη, αλλά το μέσο όρο παίρνουμε. Γι' αυτό και είπα ότι περιμένω τις προτάσεις σας. Και στο παρελθόν ε, είχαμε πολύ άριθμες τροπολογίες, οπότε περιμένω και φέτος 300 με 500. Και κατά την εξέταση των τροπολογιών θα επισέλθουμε σε όλα αυτά τα φιλεγόμενα θέματα κάτι που θα κάνουμε και στη συζήτηση των σχεδόν εισηγητών. Δεν, πάντως, ε, μακάρι να κάνετε σχετική ακρόαση για το Ρέντσι, το όχι στο δημοψήφισμα ή το ευρώ. Θα έρθω με μεγάλη χαρά να διοργανώσω τέτοια ακρόαση, αλλά είναι εκτός θέματος η σχέση με τη δική μου έκθεση όλα αυτά που είπατε. <laughs> Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ω προ το χρονοδιάγραμμα, εξέταση του σχεδίου έκθεσης σήμερα, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών, μόνο στα αγγλικά τροπολογίες παρακαλώ, ε, η διορία λήγη στι 14 Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα γίνει 25 26 Ιανουαρίου και στην Ολομέλεια κατά πάσα πιθανότητα στη δεύτερη ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε σε πιο διεξοδική συζήτηση, παρόλο που κανονικά έπρεπε και σήμερα να είχαμε επισέλθει σε λεπτομεριακή συζήτηση. Θα έχουμε ξανά την ευκαιρία τη Δευτέρα στην κοινή συζήτηση με την άλλη Επιτροπή να ξανασχοληθούμε με το θέμα. Ωραία, περνάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα που προβλέπει κοινή συζήτηση των σημείων 10, 11, 12, 13, 14 και 15 εξέταση δηλαδή των γνωμοδοτήσεων των σχέδιων γνωμοδότησης για την απαλλαγή του 2015. Ε, οι γνωμοδοτήσεις αυτές αφορούν το Γενικό Περιπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διάφορους ε, οργανισμούς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής, δηλαδή του ΣΕΝΤΕΦΟΠ, του Eurofound, ε, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Η κυρία Χάρκιν απουσιάζει, αλλά η κυρία τομό θα αναπληρώσει την κυρία Χάρκιν και θα μας ενημερώσει για τις γνωμοδοτήσεις αυτές. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους της κυρίας Χάρκη, λοιπόν, θα σας ενημερώσω για τα σημεία 10-15 της ημερήσιας διάταξης. 6 σχέδια γνωμοδότησης για την απαλλαγή του 2015. Για το Σεντεφό Eurofound EU, OSHA και ETF, το ελεκτικό συνέδριο δήλωσε ότι ε, για την διαχειριστική χρήση 2017 δεν βρέθηκαν ατασταλίες και από το Δεκέμβριο από τις 31 Δεκεμβρίου του 2015 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2015 οι λογαριασμοί ε, αντικατοπτρίζονται πιστά. Η κυρία Χάρκιν προτείνει η αναθεώρηση των σχετικών κανονισμών για, τις, για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, Eurofound και EU, EU OSA. Συγγνώμη, έχει μια δύσκολη λέξη. Ε, για την καλή διαχείριση των τριών οργανισμών. Κυρία Χάρκιν, ευχαριστεί τους συναδέλφους και την ανταλλαγή απόψεων που γίνονται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανάπτυξης των Οργανισμών, που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Χαίρεται για την ε, ενίσχυση της συστηματικής συνεργασίας ε, του ETF και του SEDEFOP. Και επίσης ε, συνεχίζεται η εφαρμογή της κοινή προσέγγισης ε, για τις αποκεντρωμένους οργανισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαιρετίζει την πρόοδο που επετέφθη κατά την ε, εφαρμογή του οδικού χάρτη. Σε ό,τι αφορά την ίδιο όσα χαιρετίζει τη συμβολή της για την προώθηση της ασφάλειας και της υγείας στον χώρο εργασίας και το σχέδιο για την περίοδο 2014-2020 και χαιρετίζει επίσης την αναθεώρηση των ε, οριακών τιμών ε, για την έκθεση των εργαζομένων στη σχετική οδηγία για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Βέβαια, δεν υπήρχε πλήρης εφαρμογή του κανονισμού 2004. Επίσης, για το Eurofund ε, χαιρετίζει τον υψηλό βαθμό εκτέλεσης, 99,9% το 2015, με καλά αποτελέσματα επίσης στο στο εργαστήριο, στο, στις εργασίες και ολοκληρώθηκαν ε, οι εκκρεμότητες με την Ιρλανδία. Σε ό,τι φορά την εφαρμογή του τρέτους προγραμματισμού, πάει καλά. Γίνονται συνεχώς πολλές μελέτες, εκδηλώσεις, σχέδια και παρουσιάσεις. Και το ΣΥΝΤΕΦΟΠ όπως και το Eurofund, έχει υψηλό επίπεδο εκτέλεση προϋπολογισμού για το 2015, 98,5% και χαιρετίζει την ποιότητα του ερευνητικού έργου του ΣΕΝΤΕΦΟΠ. Και συμφωνούμε με τις προτάσεις πολιτικής που κάνει. Η κυρία Χάρκιν επίσης θεωρεί ότι ε, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις δεξιότητες ταυτόχρονα με τις εκθέσεις αναχώρα και την ανάλυση και χαίρεται για την εγγενήση του νέου πανοράματος δεξι... δεξιοτήτων. Επίσης, ε, ε, χαίρεται για την εσωτερική ε, αναδιοργάνωση τον Ιανουάριο του 2015 ε, που συνάδει πληρώς με τον κανονισμό για το προσωπικό. 96% είναι ο συντελεστής εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο ETF, πολύ θετικό συντελεστής και τέλος οι προσπάθειες του Ιδρύματος για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια είναι πολύ θετική και ελπίζει ότι θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία στο εγγύς μέλλον. Σε ό,τι αφορά τέλος, τον, την εκτέλεση του Γενικού Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και την απαλλαγή για το 2015, θεωρεί ότι το ποσοστό φάσ, σφάλματος 5,2% που έχει διαπιστωθεί, ναι μεν ε, ε συνιστά μείωση κατά μισή ποσοστία μονάδα σχέση με πέρυσι, αλλά εξακολουθεί να είναι υψηλό. Θα πρέπει να μειωθεί το ποσοστό σφάλματος και θα πρέπει γι' αυτό τα κράτη-μέλη να στέλνουν ε, επαρκείς πληροφορίες για να αποφευθούν σφάλματα πριν ζητηθούν ε, επιστροφές ποσών. Και αν είχαν, είχε βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών, θα μπορούσε το ποσοστό σφάλματος να είναι κατά 2,4% χαμηλότερο. Επίσης, το ελεκτικό συνέδριο ε, προ συστήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την εμπειρία της προηγούμενης περίοδου 2007-2013 και να επικεντρωθεί στην ανάλυση των εθνικών κριτηρίων επιλεξιμότητας και για την επόμενη περίοδο 2014-2020 και με βάση αυτά τα κριτήρια να δίνει κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη-μέλη για την απλούστευση και αποφυγή υπερβολικά γραφειοκρατικών κανόνων. Επίση, εκφράζει την ανησυχία τη γιατί μέχρι τα τέλη του 2018 λιγότερο από το 20% των εθνικών αρμοδίων αρχών για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων είχαν ε, διοριστεί. Κάτι που σημαίνει ε, μεγάλο κίνδυνο καθυστέρηση τη εκτέλεση για το πρόγραμμα 2014-2020, τη σχετική δηλαδή δημοσιονομική περίοδο. Thank uh, uh, Σας ευχαριστούμε για αυτή την ε, παρέμβαση και καθότι είμαστε τόσο λίγοι αυτή τη στιγμή στην αίθουσα, θα σας διαβάσω απλώς το χρονοδιάγραμμα των εργασιών. Η προθεσμία λοιπόν για την υποβολή τροπολογίων είναι η 14η Δεκεμβρίου στις 12 ε, το μεσημέρι, 25 Ιανουαρίου, υιοθέτηση στην Επιτροπή 22 και 23 Μαρτίου μετά η ψηφοφορία στην της ουσίας αρμόδια επιτροπή και τέλος η ψήφιση στην Ολομέλεια στα τέλη Απριλίου, 26-27 Απριλίου. Ε, Θα δώσω το λόγο στην κυρία Χέλγα Στίβανσον που ήθελε να πάρει το λόγο σε σχέση με αυτό το σημείο τη ένταξη. ένταξης. Παρακαλώ λοιπόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώμη για τη σύγχυση. Ε, σας διαβάζω λοιπόν αυτήν τη δήλωση εκ μέρους του αδερφού Μπασίρου, ο οποίος δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα εδώ. Δηλώνω, λοιπόν τα εξή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την ε, για, ε, για αυτή την ε, πρόταση και ε, ο ποσοστό σφαλμάτων στον τομέα της απασχόλησης έχει μειωθεί ειδικότερα σε σύγκριση με την απαλλαγή του προπολισμού για το 2014. Παρόλα αυτά, θεωρώ πως αυτό το ποσοστό ε, παραμένει υπερβολικά υψηλό ε, και σχετίζεται και με μια σειρά από περαιτέρω στοιχεία στην αξιολόγηση από την πλευρά του Ελεκτρικού Συνοδρίου. Και όπως ε, αναφέρει σωστά και η κυρία Χάρκιν, υπάρχουν κίνδυνοι ε, για την καθυστερημένη εκτέλεση του σημερινού προπολογισμού που το Ελεκτικό Συνέδριο φοβάται πολύ ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερος από αυτές τι τελευταία προγραμματικής περίοδου. Κάτω Τέλο τη τελευταία ε, προγραμματική ε, περίοδου είχε γίνει πολλή λόγο για την αποφυγή των καθυστερήσεων και η δική μα λοιπόν πολιτική ομάδα διαπιστώνει με μεγάλη ανησυχία ότι η κατάσταση αντί να βελτιωθεί επιδεινώθηκε. Υποστηρίζουμε την έκκληση που κάνει το ελεγκτικό συνέδριο να για την επανεξέταση από την πλευρά τη Επιτροπής ε, των μηχανισμών εκτέλεση των διαρθρωτικών ταμείων στο μέλλον ε, και σε ό,τι αφορά την ε, θέσπιση απλουστευτικών μέτρων. Επίσης, ε, το ΙΣΑ υποστηρίζει τα μέτρα που επιτρέπουν μια πιο στοχευμένη πολιτική και τα όσα προτείνει το ελεγκτικό συνέδριο σε ό,τι αφορά την καλύτερη αξιολόγηση των τρέχοντων προγραμμάτων. Θα θέλαμε να υποστηρίξουμε περαιτέρω μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση και σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες, το ECR εδώ και πολύ καιρό θεωρεί ότι υπάρχουν μεγάλες ανεπάρκειες στο σύστημα ε, της χρηματοδότησης των υπηρεσιών και ε, εδώ θα υπήρχαν πολύ ε, μεγάλες δυνατότητες για εξοικονομήσεις κονδυλίων στο πλαίσιο του προπολογισμού. Ακτιμούμε τις προσπάθειες που έχουν κάνει οι εν λόγω υπηρεσίες, ούτως ώστε να συντονίσουν τις εργασίες τους και να αποφύγουν την επικάλυψη των εργασιών τους. Ωστόσο, θεωρούμε πως θα πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες. Ευχαριστούμε θερμά την ε, κυρία Χάρτιν για το ε, έγγραφο, αλλά θα υποβάλουμε και κάποιες ε, τροπολογίες σε σχέση με τα ζητήματα που μόλις τώρα έθιξα και αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την συνεργασία με τους ε, συναδέλφους. Αυτή ήταν η δήλωση λοιπόν εκ μέρους του κυρίου Μπασίρ, την οποία μόλις τώρα σε διάβασα. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος, η ε, κυρία Στίβενς, που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Δυστυχώς, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει μεγάλη απαρτία σήμερα στην αίθουσα. Θα πρότεινα λοιπόν να σταματήσουμε εδώ την συνεδρίασή μας. Υπάρχει ένα ακόμα σημείο στην ημερήσια διάταξη, τον οποίο νομίζω πως δεν έχει νόημα να συζητήσουμε. δεν έχει νόημα να έχουμε ένα τέτοιο θέμα στην ημέρησια διάταξη όταν έχουμε τόσο λίγους συναδέλφους στην αίθουσα. Εσείς βέβαια είστε οι συντάκτε της ομοδότησης, για αυτό το σημείο κυρία Στίβενς, αλλά από εσά λοιπόν εξαρτάται. Θέλετε τώρα να αναφερθείτε σε αυτή τη γνωμοδότηση ή θέλετε να περιμένετε όταν θα έχουμε περισσότερους συναδέλφους εδώ παρόντες. Καλώς συμφωνείτε μαζί μου, οπότε θα περιμένουμε για να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα την επόμενη φορά που θα έχουμε περισσότερους συναδέλφους εδώ στην αίθουσα. Η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι η 14η Δεκεμβρίου, αλλά η ψηφοφορία δεν θα λάβει το σε άλλος χώρα έως τα τέλη Ιανουαρίου. Δεν νομίζω λοιπόν πως έχει νόημα με μόνο τρία μέλη της Επιτροπής παρόντα να μένουμε στην αίθουσα και να συνεχίσουμε αυτή τη συνεδρία. Please. Uh, thank you, Chair. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αντιλαμβάνομαι πλήρω τι ανησυχίε που εκφράσατε σε ό,τι αφορά την απουσία των συναδέλφων από την αίθουσα. Ε, Ενδεχομένω θα έπρεπε να επανεξετάσουμε την προθεσμία υποβολή τροπολογιών που είναι η 14η ε, Δεκεμβρίου, δηλαδή την ε, επόμενη εβδομάδα. Κατά συνέπεια δεν θα έχω τη δυνατότητα να πάρω το λόγο για αυτό το ζήτημα. Οπότε, αν μου επιτρέπετε, εγώ θα ήθελα να κάνω μια επανέμβαση. Μπορώ να το κάνω πρόεδρε. Καλώς σας, ευχαριστώ. So this is regarding the Marrakesh. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία του Μαρακές. Broadly supported by... Θα ήθελα να ε, υποστηρίξω την ε, συμφωνία από την πλευρά τη Επιτροπή ε, που έχει λάβει την υποστήριξη όλων των ατόμων με την αναπηρία δικότερα τη Ένωση Τυφλών και θα ήθελα να ασκήσουμε πιέσεις ούτως ώστε να υιοθετηθεί το ταχύτερο δυνατό αυτή η ε, συμφωνία. Θα πρέπει δηλαδή να σταματήσει το ταχύτερο δυνατό η πείνα, ο λοιμό, αν θέλετε, ε, σε ό,τι αφορά την ανάγνωση βιβλίων για ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα όρασης. Ούτως ή άλλως αυτό το δικαίωμα είναι κατοχυρωμένο στις συνθήκες της Ένωσης, αλλά από εκεί και μετά έχουμε και την ηθική υποχρέωση να παρέχουμε πρόσβαση σε όλους σε βιβλία. Δεν είναι μόνο θεμελιώδου σημασία για τη μόρφωση, αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικά για, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια εικόνα για τον κόσμο. Η δική μου λοιπόν γνωμοδότηση ακολουθεί ουσιαστικά την συμφωνία LPD και τη συμφωνία του Μαρακέ. Για παράδειγμα, στο σημείο 7 γίνεται αναφορά στην πρόσβαση στι πληροφορίε. Το CRPD όμω αναφέρει ότι πρόκειται για πρόσβαση σε πληροφορίε και στην επικοινωνία. Οπότε εμεί με την δική μα ε, ε, γνωμοδότηση κάνουμε αυτή τη διόρθωση. Επίση, θεώρησα σημαντικό ε, να συμπεριλάβουμε εδώ τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν άλλα προβλήματα εκμάθηση, όχι δηλαδή μόνο τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα δυσλεξία σε σχέση με την ανάγνωση ενό βιβλίου στην παραδοσιακή του μορφή. Επίση, με περαιτέρω ε, τροπολογίες ε, θέλησα να διασφαλίσω ότι όλε οι πληροφορίε, δηλαδή και επιγραμμικέ ε, και μη επιγραμμικέ, θα πρέπει να είναι διαθέσιμε, γνωρίζοντα ότι και λαμβάνοντα υπόψη ότι η γνώση ω τέτοια ταχύ, εξελίσσεται ταχύτερα από την νομοθεσία και δεν ξέρουμε ποιε άλλε μορφέ διαβίβασή τη. θα ε, προκύψουν στο μέλλον. Επίσης ε, θεωρώ ε, πολύ σημαντικό το να λάβουμε υπόψη μας τις απόψεις των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία στην έκθεση της Επιτροπής η οποία θα υποβληθεί σε πέντε χρόνια. σε ό,τι αφορά την οδηγία 2001. Ή μάλλον η παρέμβαση που έκανα μέχρι τώρα αφορά του σχετικού κανονισμού, Τώρα θα αναφερθώ στην οδηγία. Οι ε, τροποποιήσεις λοιπόν που προτείνω σε σχέση με την οδηγία ακολουθούν το ίδιο πνεύμα με αυτές ε, που ανέφερα μόλις τώρα σε σχέση με τον κανονισμό. Δηλαδή περιεχόμενο τόσο επιγραμμικό όσο και μη επιγραμμικό θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και επίση, με βάση τον ορισμό τη συμφωνία ε, του Μαρακέ, ε, διευρύνω τον ορισμό των ατόμων που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία για να συμπεριλάβω τα άτομα εκείνα με αναπηρία τα οποία δεν έχουν την δυνατότητα να ε, κρατήσουν στα χέρια τους ή με άλλο τρόπο να μεταχειριστούν ένα βιβλίο. Σημειώνω επίσης ότι ο χάρτης των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων απαγορεύει τις διακρίσεις ε, με βάση την αναπηρία και θεωρώ πως αυτό είναι σημαντικό να τονιστεί ακόμα περισσότερο εδώ. Επίσης θεώρησα πολύ σημαντικό και εδώ να συμπεριληφθεί ο ρόλος ε, των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία ε, και ειδικότερα ένας των τυφλών συμφωνεί ιδιαίτερα με τις δικές μου προτάσεις και ελπίζω ότι θα μπορέσετε να υποστηρίξετε την προσέγγιση και τις πρότασεις που σας έκανα εδώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Εμείς σας ευχαριστούμε που ήρθατε λέει Πρόεδρος. Ευχαριστούμε για τη δουλειά σας, αλλά δεν έχουμε, από ό,τι φαίνεται. να αλλάξουμε την πρόθεσμη για τις τροπολογίες, άρα παραμένει 14-12 και θα εγκρίνουμε το κείμενο 25-26 Ιανουαρίου στην ε, Επιτροπή μας και θα ψηφίσει η κυρίως αρμόδια Επιτροπή, η Νομική Επιτροπή, την 31η Ιανουαρίου. Επομένως, εδώ ολοκληρώνεται η συνεδρίασή μας. Και είμαι βεβαία ότι θα επανέλθουμε κατά κάποιο τρόπο όσον αφορά τα θέματα από 10 έως 15. Θα γίνει αυτό ένα τμήμα της συζήτησης που θα έχουμε στο Στρασβούργο έχουμε αυτή την κοινή συνδέση με την Οικονομική Επιτροπή, οπότε θα υπάρξει ευκαιρία να υποβληθούν ερωτήσεις. Για όλα τα θέματα αυτά τα οποία δεν μπορέσαμε να δουλέψουμε, μια που συνάδελφοι είναι σε άλλες συνεδριάσεις και δεν μπορούσαν να έρθουν, οπότε θα τα ξαναπούμε. Sorry, I think we must. Uh, uh, uh, it's no good order to work like this. My proposal is. Όχι, δεν ωφελεί να δουλεύουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Οπότε σας προτείνω να ευχαριστήσουμε την κυρία Στέφανης για τη δουλειά της. Και για τα σημεία 10-15 να συζητήσουμε στη συνεδρίαση στο Στρασβούργο την άλλη εβδομάδα την επομένη. Σας ευχαριστώ που ήρθατε.